E Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Ρούμπιχ. Ε, επί διαδικαστικού. Κύριε Ρούμπιχ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΣΤΟΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας παρουσιάσω τον κύριο Τιφ Τόλον που είναι ε, επικεφαλής του προγράμματος στη Ζάμπια. Θα ήθελα να τον συγχαρώ γιατί πήρε το βραβείο ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να τον χαιρετήσουμε εδώ από, το, από τα έδρανα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούμπιχ. Ε, Βεβαίω και ε, η Προεδρία συγχαίρει και συγχειροκροτεί με την αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο, στην κυρία Μοργάντη. Μοργάντη, παρακαλώ κύριε Μοργάντη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ε, στην ε, μνήμη των ε, θυμάτων του κρουαζιερόπλου Κώστα Κονκόρδια στα ανοιχτά του Ισενίσου Τζίλιο. Είναι 11 τα πιστοποιημένα θύματα διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα 29 αγνοούμενοι. Επομένως θα μπορούσε να γίνει είναι ακόμα χειρότερος ο απολογισμός, βαρύτερος πρόεδρος. Η Προεδρία και όλοι οι συναδελφοί βεβαίως εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και λύπη για τα όσα συνέβησαν. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.